Στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής που στη συζήτηση θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Λεσκεβίτσιους, τον εκπρόσωπο της Λιθουανικής Προεδρίας. Ο κ. Λεσκεβίτσιους είναι Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Λιθουανίας. Η δήλωση αφορά τις εξαγωγές όπλων και την εφαρμογή της κοινή θέσης του Συμβουλίου. Ακούμε πρώτα τη δήλωση του Υπουργού. Για πέντε λεπτά. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για το θέμα της υλοποίησης της κοινή θέσης από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τρέχουσα ε, άποψη της ε, αντιπρόεδρο τη Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου. Οι κοινέ θέσει είναι από τα πιο αναπτυγμένα εργαλεία ε, στον τομέα της εναρμονισμένων εξαγωγών όπλων. Ξεκινά από τον ε, κώδικα διοντολογίας που είναι δεσμευτικό δεσμευτικό κείμενο και εκεί κύριος στόχος είναι να κάνει τις εξαγωγές πιο υπεύθυνε. Και το κάνει αυτό απαιτώντα ότι οι εξαγωγέ όπλων από τα ευρωπαϊκά μέλη θα πρέπει να ελέγχονται και να εξουσιοδοτούνται πριν από την μεταφορά των όπλων στο εξωτερικό. Και αναφέρεται και σε εξαγωγέ σε τρίτε χώρε ε, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινή θέση, τα κράτη-μέλη απαιτείται να αξιολογήσουν οποιασδήποτε εξαγωγές όπλων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση κάποιες παραμέτρους που περιλαμβάνουν τον ε, κίνδυνο ε, να δημιουργήσουν παραβίαση ε, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το, ο κίνδυνος επίσης ε, να φτάσουν αυτά τα όπλα σε ε, χρήστες στο οποίους δεν προορίζονται και την ε, όξυνση συγκρούσεων. Ταυτόχρονα ορίζει η θέση ότι κάθε αίτηση θα πρέπει να αξιολογείται μία-μία ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι θέματα όπως ε, οι τελικοί χρήστες, η ποιότητα των όπλων, οι περιστάσεις από τις οποίες ε, γίνεται η εξαγωγή, όλοι αυτοί είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης, ε, υπονοεί το γεγονός ότι κάποια εξαγωγή προς μια συγκεκριμένη χώρα δεν σημαίνει ότι μια συγκεκριμένη χώρα είναι ή πρέπει να είναι υπό εμπάργο όπλων. Ορίζοντας αυτά τα κριτήρια, ε, κάποιοι μηχανισμοί διαβούλευσης, επίσης ε, η κοινή θέση εναρμονίζει ε, τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών και αυτός ο στόχος περιορίζεται με την, τον μηχανισμό απόρριψης εξαγωγών και πρέπει να υποβάλλεται κάποια συγκεκριμένη αίτηση τα κράτη-μέλη ανταλλάσσουν απόψεις για τις εξοργές όπλων και τις ε, πολιτικές. Ε, η ομάδα ε, εργασίας για την επεξεργασία των εξαγωγών σημαντικών όπλων, η άρμα ασχολείται με αυτά τα θέματα στο Συμβούλιο. Θα έχει επίσης διατάξεις σχετικά με την υλοποίηση που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της λειτουργίας. Ε, θα πρέπει να δούμε το κοινό πλαίσιο που ε, αφορά και τα 28 κράτη-μέλη για όλες τις εκλογές όπλων σε εθνικό επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές. Άρα η εξόλυση κινδύνου που γίνεται από ένα κράτος μέλος μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι η κοινή θέση καθορίζει μια υποχρέωση διαδικασίας αλλά όχι αποτελέσματος για το κράτος μέλος που κάνει την αξιολόγηση κινδύνου των αιτήσεων εξαγωγών. Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν μελετάμε τις υποχρεώσει που επιβάλλει κοινή θέση στα κράτη-μέλη και ε, πρέπει να αναφερθούμε στις πιθανές παραβιάσεις. Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να είναι υπόλογα ε, στις αποφάσεις εξαγωγών όπλων, χάρη στο γεγονός ότι η κοινή θέση περιέχει ε, μια διάταξη για την διαφάνεια. Επίσης, ε, απαιτείται ε, να δημοσιεύονται λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις για τις εξαγωγές των όπλων. Αυτές οι εκθέσεις ε, θα πρέπει να πληρούν τα ύψιστα πρότυπα σε ό,τι αφορά τα, τις εξαγωγές όπλων. Η διαφάνεια είναι προαπαιτούμενα και ένα μεγάλο, σημαντικό μέσο για την πολιτεία των των πολιτών για να ασκούν τον δημοκρατικό έλεγχο ε, στις κυβερνητικές αποφάσεις για τις εξαγωγές όπλων. Θα ήθελα τώρα να πω ε, μερικά λόγια για την αναφερετική διαδικασία της, ε, που έλαβε χώρα. Wow. Η αναθεώρηση ξεκίνησε στις αρχές του 2012 μετά από μια ενδελεχή ανάλυση των απαντήσεων σε ένα αναλυτικό ρευματολόγιο. Τα, αναλυτικά, τα Προκαταρκτικά αποτελέσματα αναφέρονται στα πορίσματα του Συμβουλίου στις 19 Νοεμβρίου 2012 και επιβεβαιώνουν πόσο καλό είναι το κείμενο της κοινή θέση, αλλά τόνισαν ότι χρειάζεται και περαιτέρω εργασία για την εφαρμογή των διατάξεών του. Η ομάδα εργασία του Συμβουλίου προσπαθεί να βελτιώσει διάφορε πλευρέ εφαρμογή τη κοινή σε συμπεριλαμβανομένη τη ε, ανταλλαγή πληροφοριών για τον τελικό στόχο και την ε, ε, ανταλλαγή ενημερώσεων. Στόχος μας είναι να αυξηθεί ο, όγκο όγκος και η αξία των πληροφοριών που ανταλλάσσουμε με πιο ε, χρήσιμη, πιο σχετική και πιο έγκαιρη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Αυτέ οι βελτιώσεις θα έχουν ε, ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί ο χρήστη, ο, συγγνώμη, το εγχειρίδιο χρηστών που θα μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε και να εφαρμόσουμε την κοινή θέση. Το Κοινοβούλιο και η Κοινωνία των Πολιτών ε, ενημερώνονται για τα διάφορα στάδια της αναθεώρησης μέσω μια συνάντηση με τι σχετικέ μη κάπα όμικρον ανά εξάμεινο και των παρουσιάσεων που κάνουμε στην υποεπιτροπή σα για την ασφάλεια και την άμυνα. Υπενθυμίζω ότι η κοινή θέση εφαρμόζεται και μια σειρά από χώρες. χώρε. Επίση, θέλουμε αυτά τα κριτήρια και η διαφάνεια που αναφέρεται στην κοινή θέση να εφαρμόζονται και από τρίτε χώρε με ένα ε, φιλόδοξο πρόγραμμα και με την τελευταία μας απόφαση που πήραμε τον Νοέμβριο του 2012 να διαθέσουμε 1,8 εκατομμύρια για αυτό το σκοπό. Τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στις πρώτες γραμμές της βελτίωσης της παγκόσμιας ε, διαδικασίας ελέγχου των ε, εξαγωγών όπλων μέσω των διαπραγματεύσεων που γίνονται στα Ηνωμένα Έθνη για την συμφωνία για τις εξαγωγές όπλων. Το 2013 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε αυτήν την συνθήκη και είναι η πιο φιλόδοξη προσπάθεια ρύθμισης των εξαγών όπλων. Επιτρέπει περισσότερη διαφάνεια που θα εφαρμοστούν από όλα τα κράτη-μέλη που θα την εφαρμόσουν. Αυτή η συνθήκη για το εμπόριο όπλων θα συμβάλλει στην ειρήνη και την ασφάλεια και την μείωση των δεινών και της βίας. Για να αρχίσει να ισχύει πρέπει να επικυρωθεί αυτή η συνθήκη τουλάχιστον από 50 κράτη-μέλη των ΗΠΑ. Ε, τα κράτη-μέλη της Ένωσης εξέφρασαν την επιθυμία τους να επικυρώσουν ταχαίως την συνθήκη και εσείς ε, κύριοι ευρωβουλευτές παίζετε ρόλο γι' αυτό. Επειδή καλύπτει αυτή η συνθήκη κάποιους τομείς νέας αρμοδιότητας ή σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ζητηθεί πριν ε, ε, επιτρέψει το Συμβούλιο την επικύρωση από τα κράτη-μέλη. Βασιζόμαστε στη στήριξή σα, ούτω ώστε αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί τάχιστα και να υπάρξει η κρίσιμη μάζα των 28 κρατών μελών, ούτω ώστε να φτάσουμε γρήγορα τα 50 που απαιτούνται για το όριο εφαρμογής της νέας Συνθήκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λεσκεβιτσούτ. Ο κύριος Γκάλερ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τα όπλα δεν είναι συνηθισμένο εμπόρευμα. Αν πέσουν σε λάθος χέρια, κάνουν ζημιά. Εάν όμω είναι υπό τον έλεγχο υπευθύνων κυβερνήσεων, μπορούν να παίζουν αποτρεπτικό ρόλο, να εμποδίζουν συγκρούσει και μπορούν να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά κράτη και να οδηγήσουν και ε, στην αποκατάσταση των δικαιωμάτων των λαών. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι καλό ότι από κοινού έχουμε μια διαδικασία για την έγκριση στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμών. Αυτό που επιδιώκουμε δεν το έχει επιδιώξει καμία άλλη κοινότητα κρατών και φαίνεται πως είναι τόσο καλή η προσπάθειά μας που και τρίτες χώρες χρησιμοποιούν τους κανόνες μας, εφαρμόζουν τους κανόνες μας. Η κοινή θέση από το Μάρτιο 2008 είναι ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο με οκτώ διατάξεις και όπως ξέρετε εκπονήθηκε και ένας, ένα εγχειρίδιο χρήσης με βάση τα κριτήρια αυτά. Διαπιστώνουμε ότι φυσικά εμείς ως Κοινοβούλιο ε, δεν έχουμε ε, δυνατότητα συναπόφασης. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την ερμηνεία σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αίτηση εξαγωγή. Αλλά οι εθνικοί μας συνάδελφοι έχουν συγκεκριμένο ρόλο να φροντίσουν ούτω ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να ελέγχονται οι κυβερνήσει τους να εφαρμόζουν σωστά αυτές τις κοινέ προδιαγραφές που περιέχονται στην κοινή θέση. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν συνέπεια σε επίπεδο ένωσης και αυτό είναι το καθήκον μας με βάση και την ηγεσία της κυρίας ε, Άστον και εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε να ενημερωνόμεθα τακτικά. Υποστηρίζουμε ως ε, πολιτική ομάδα και τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων και ελπίζουμε να αρχίσει να εφαρμόζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκαλέρ. Κύριε Κοπά, ένα λεπτό. Το ζήτημα της σωστής εφαρμογής της κοινή θέση για την εξαγωγή όπλων δεν είναι τεχνικό είναι ζήτημα ύψιστης της πολιτικής σημασίας που αφορά το κατά πόσο θέλουμε να είμαστε στην πραγματικότητα συνεπεί στις δεσμεύσεις μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. είναι λοιπόν ντροπή το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα με την λίγο πολύ σιωπηρή υποστήριξη των συντηρητικών και φιλελεύθερων οδήγησαν στην καταψήφιση της σχετικής έκθεσης πρωτοβουλία της συναδέλφου lsing στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων. τώρα παρουσιάζουν κοινή πρόταση ψηφίσματος που δεν αναφέρει κανένα σχεδόν από τα ουσιαστικά προβλήματα. η αλήθεια είναι ότι δεν επιθυμούν πραγματικό έλεγχο στην εξαγωγή όπλων και εδώ είναι η διαφορά μας. εμείς επιμένουμε και τονίζουμε ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές την ανάγκη να σταματήσει η υποκρισία εκ μέρους των μεγάλων κατασκευαστών όπλων να υπάρξει διαφάνεια και έμπρακτη εφαρμογή της απαγόρευσης εξαγωγής σε δικτατορικά κράτη και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει βάσιμη υποψία ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταστολή ελευθεριών και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. σας ευχαριστώ. Κυρία Κοπά, κάρτα. Ευρωβουλευτή. Σας εκτιμώ ιδιαίτερος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θυμάστε ότι στη συνεδρίαση της ΑΦΕΤ, γιατί αναφερθήκατε στο σχέδιο έκθεσης της κυρίας Λέζινγκ, σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι η ψηφοφορία είχε το εξή αποτέλεσμα. Κανεί κανείς δεν ε, ψήφισε υπέρ ε, και μία αποχή είχαμε, ενώ οι υπόλοιπε ομάδες ψήφισαν κατά της έκθεσης Λέζινγκ αγαπητέ συνάδελφε αν θυμάστε καλά αποσύρατε την υποστήριξή σας από μια έκθεση στην οποία είχαμε σχεδόν συμφωνήσει. λοιπόν όλοι εδώ μέσα έχουμε μνήμη όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει. μην ανοίξουμε μερικά θέματα που δεν συμφέρουν κανένα. Ευχαριστώ. Έκλεισε το θέμα. κυρία Νικολάη. Δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε καλύτερη και ουσιαστική εφαρμογή της κοινή θέση με βιώσιμο όμως τρόπο και αμοιβαίως ε, επωφελή και για τη βιομηχανία και για αυτούς που, θέλει να προστατεύσει. Μερικές προτάσεις κατά τη γνώμη μας είναι ουτοπικές γιατί θα πρέπει να έχουμε κάποιες εγγυήσει για όλα τα κράτη-μέλη ότι ε, καμία παρα, παραστρατιωτική οργάνωση ή μη κυβερνητική δομή δεν βρίσκεται πίσω από, μια, από ένα συμβόλαιο αγοράς. Δεν θα πρέπει επίσης να οδηγήσουμε σε ασφυξία την αμυντική βιομηχανία, να αποφύγουμε οποιαδήποτε ριζοσπαστική προσέγγιση και να προωθήσουμε καλύτερη συνεργασία για την κοινή θέση προκειμένου να μπορέσει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας να προωθήσει την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ του ελέγχου των όπλων και την πρόθεση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία. Ε, η λύση είναι η πραγματική ολοκλήρωση και εμπέδωση της βιομηχανίας μας. Σε ό,τι αφορά την συμβαστική λύση για την κοινή θέση, αυτή είναι σημαντικό βήμα πρόοδου και θα πρέπει να, είναι, να είμαστε ρεαλιστικοί πριν ε, διεκδικήσουμε περισσότερα. Ευχαριστώ κυρία Κρόνμπερκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ είναι μια ξεχωριστή κατάσταση. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια κοινή θέση για τι εξαγωγέ των όπλων, που είναι μοναδική συμφωνία και ένα πολιτικό εργαλείο το οποίο καθορίζει σαφή κριτήρια για το εμπόριο των όπλων. Φέτο και ο ΟΗΕ ε, ενέκρινε την συνθήκη για το εμπόριο των όγκρων. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, πιο προοδευτική πολιτική στον τομέα αυτό. Υπάρχουν δύο ψηφίσματα που είναι έτοιμα προς ψήφιση. Το ένα από τους σοσιαλιστές, του πράσινου και την ΚΟΕ αυτό το ψήφισμα ε, είναι για να βελτιώσει την κοινή θέση σε θέματα όπως είναι η διαφθορά, η διαφάνεια και η συνέπεια εφαρμογής ε, των κοινών κριτηρίων των κρατών μελών. Το δεύτερο ψήφισμα από τον ΑΛΔΕ, το ΕΛΚ και το ECR θεωρεί αρκετά καλή την κοινή θέση και δεν την ε, προωθεί σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Θεωρεί ότι είναι ένα βήμα προς τα πίσω σε σχέση με την κοινή θέση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα ότι το ψήφισμα αυτό είναι έσχυντο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων δικαιωμάτων είναι η προσθέμενη αξία της κοινή θέση. Είναι σημαντικό ιδιαίτερα ε, δεδομένη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική όπου κατευθύνονται ε, τα, οι όπλων. Εκεί ε, στο ψήφισμα αυτό του ΕΛ και του ΕΛ του ε, δεν υπάρχει αναφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ψηφοφορία αύριο θα δείξει προς ποια πλευρά τίθεστε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει κύριος Βλάσακ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να πω επ' ευκαιρία του θέματος ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι εξαγωγείς ε, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που, δεν, ε, που είναι εγκλωβισμένες όπως η Τσεχία, η Πολωνία, η Γερμανία, και, ε, μάλλον η Τσεχία που θα πρέπει να περάσουν από τα λιμάνια άλλων χωρών, Γερμανίας, Πολωνίας, κάτι που προϋποθέτει επιπλέον έγκριση και έτσι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το θέμα της άδειας από τη χώρα προέλευσης. Το βήμα αυτό έχει πολιτικό υπόβαθρο και πολλές φορές καθυστερεί την όλη διαδικασία και μερικές φορές οδηγεί και σε πλήρη απόρριψη της άδειας. Κάτι που επαυξάνει το κόστος με αποτέλεσμα να χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους οι βιομηχανίες μας και να υφίστανται τεράστιες οικονομικές ζημιές γιατί είναι ένας κλάδος με τεράστια προστιθέμενη αξία που εξασφαλίζει δεκάδες χιλιάδες θέσεων απασχόλησης και δεν θα πρέπει να καταβαραθρωθεί. Είναι απαράδεκτο χώρες όπως η Τσεχία να βρίσκονται σε διακριτική μεταχείριση και να υφίστανται τη δυσμενή ε, μεταχείριση εξαιτία αυτή τη συμφωνία για τι εξαγωγέ. Θα ήθελα να ζητήσω από τι αρμόδιε αρχέ να ελέγξουν το κατά πόσο απαιτούνται αυτέ οι επιπρόσθετε άδειε ή εγκρίσει, κατά πόσο ένα τέτοιο μέτρο είναι ανάλογο με το σκοπό που επιζητούμε και κατά πόσο το, η προπόθεση αυτή συνάδει με το άρθρο 36 τη συνθήκη. Κοιτάξτε, στο Μάλι οι ε, αντάρτες πυροβολούν με γερμανικά όπλα κατά των Γάλλων και Γερμανών στρατιώτων. Η Γερμανία στέλνει στρατιώτες ε, να υποστηρίξουν ε, τα στρατεύματα στο Κατάρ. Η, όπως σας είπα και στο Μαλί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Πρέπει να απαγορευτούν αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρουμε τι συμβαίνει όταν ε, ε, η τεχνολογία, η στρατιωτική και τα όπλα δίδονται σε αυταρχικά καθεστώτα. Ξέρουμε ότι τα χρησιμοποιούν για να δολοφονούν ανθρώπους, για να κάνουν βασανιστήρια. Ξέρουμε ότι ε, θα πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Και γι' αυτό αποφασίστηκε αυτή η κοινή θέση για την, τον έλεγχο των εξαγωγών των όπλων. Αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει αποτέλεσμα και δεν είναι πρόκειτο να λειτουργήσει γιατί είναι χρήσιμα για τα κέρδη της βιομηχανίας όπλων και είναι χρήσιμο για να έχουμε και χρήσιμους εταίρους για στρατηγικούς στόχους. Έτσι έχει δώσει όπλα η Γερμανίδα Καγκελάριος στη Σαουδική Αραβία και θα παραμείνει η κατάσταση. Γι' αυτό απέρριψε η συμπληρωτική πλειοψηφία την έκθεσή μου γιατί είχα στόχο να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η κοινή θέση. Είχα κάνει προτάσεις που έχουν πολύ ευρύ απήχηση στην κοινωνία των πολιτών, αλλά και από επίσημες χριστιανικές οργανώσεις. Επίσης, αυτό λέω προς εκείνους που εδώ σε αυτό το σώμα λένε ότι είναι χριστιανοί και που λένε ότι θέλουν να είναι παράγον η ειρήνη στην Ευρώπη. Όποιος θέλει να είναι παράγον ειρήνη στην Ευρώπη μπορεί να το κάνει αύριο πρέπει να ψηφίσει για το κοινό ψήφισμα των Πρασίνων, Σοσιαλδημοκρατών και της Γκουε που αναφέρει σημαντικά σημεία της απορριφθήσης εκθέσεώς μου και καλύπτει όλα τα ζητήματα. Και για την ερώτηση του κυρίου Λίζε θέλω να απαντήσω. Η συντηρητική πλειοψηφία ε, ε άλλαξε τόσο πολύ την έκθεσή μου που μπορούσαμε μόνο να την καταψηφίσουμε. Και τότε είπαν εκείνοι ότι θα ήθελαν να την ε, υπερψηφίσουν. Μα τι έννοια έχει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Λέζινγκ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Αλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον έλεγχο των εξαγωγών όπλων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο ήδη από το 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε τον κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων, καθορίζοντας οκτώ κριτήρια για τις εξαγωγές αυτές. Τα τελευταία χρόνια είναι συνεχείς οι προσπάθειες για την ενίσχυση και εναρμόνιση των πολιτικών των κρατών μελών στο θέμα της εξαγωγής όπλων. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική είναι μια κρίσιμη δοκιμασία για τις κυβερνήσεις για να αποδείξουν ότι παίρνουν στα σοβαρά την εφαρμογή μιας συνθήκης που βάζει τον άνθρωπο και την ασφάλειά του ως προτεραιότητες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τον εξοπλισμό χωρών με όπλα, ειδικότερα σε σχέση με την Συρία, όπου η κατάσταση επιδεινώνεται, οι αποφάσεις για την αποστολή όπλων εκεί και αλλού θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της συνθήκης. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος τα όπλα που παρέχονται σε ομάδες να χρησιμοποιηθούν και να διαπραχθούν άλλες πράξεις κυρία πρόεδρε το δικό μου όνειρο ήταν να μην υπάρχουν όπλα. εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι όπου γίνονται σειράξεις τα πιο σύγχρονα όπλα υπάρχουν και στις πιο ακραίες ομάδες. ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαλαβράκο. Το λόγο έχει ο κύριος Λίζεκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, φυσικά όλοι θα θέλαμε να ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο επικρατεί η ειρήνη, κανένας ε, δεν πολεμάει εναντίον κανενός, ε, σε έναν κόσμο χωρίς όπλα. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, ε, αλλά δυστυχώς δεν ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο. Οπότε στο σημερινό κόσμο δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει de facto το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό σύστημα και αν προηγουμένως σε, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό σύστημα του ελέγχου των εξαγωγών τέτοιο καλό σύστημα αποτελεσματικό ελέγχου των εξαγωγών δεν έχουν ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε κανένα άλλο μεγάλο παραγωγό όπλο στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπόδειγμα προ μίμηση για άλλε χώρε ό,τι αφορά τι εξαγωγέ, τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων. Και θα ήθελα να πω στην κυρία Λέζινγκ ότι πιστεύω ότι ο έλεγχο αυτό σήμερα ε, είναι αποτελεσματικό, λειτουργεί και επαρκεί κιόλα η Ευρωπαϊκή Ένωση και κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έκανε εξαγωγές ε, σε χώρες στις οποίες επικρατούσε εμπόλεμη σύραξη και αυτή ήταν θεμελιώδης αρχή που τήρησαν όλες οι αρχές ε, και όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα οι χώρες που παράγουν όπλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε και στην διαμόρφωση παγκόσμιων προδιαγραφών, γιατί εμείς ξεκινήσαμε με την ε, συνθήκη για το εμπόριο όπλων που έγινε δεκτό στον ΟΗΕ στις ε, αρχές του έτους. Εμείς λοιπόν δώσαμε και πάλι το πρώτο το καλό παράδειγμα. Και φυσικά θέλουμε να συμβάλλουμε στην ειρήνη του, του κόσμου, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι κοινή επιθυμία και κοινό στόχος για όλους μας. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη να εμποδίσει το εμπόριο όπλων που ε, υποδαβλίζει ε, ε, σειράξει στις διάφορες περιοχές του κόσμου και να βοηθήσει δικτατορίες να καταπιέζουν τους πολίτες τους. Γι' αυτό και έχουμε την υποχρέωση και το καθήκον να ελέγχουμε σχολαστικά τον τελικό προορισμό των τεχνολογιών και των όπλων που παράγονται στην Ευρώπη και μεταφέρονται μέσω ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί δεν γίνεται τέτοιο έλεγχο από τα κράτη-μέλη. Και αυτό τον έργο προσπαθεί να εμποδίσει η δεξιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσουμε, γιατί με τέτοιε πολιτικέ ε, εκδημοκρατισμού και ε, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να γίνονται θυσία στις ε, προσπάθειες για τις εξαγωγές όπλων. Ζητούμε διαφάνεια όλων των πληροφοριών που αφορούν τις εξαγωγές, μεταφορές, τεχνολογίες, πολεμικής και όπλων προς τρίτες χώρες και ιδιαίτερα σε περιοχές με εμπόλεμες σειράξεις. Επίσης ε, θα πρέπει να εφαρμόζεται έλεγχος ε, από όποιες διάβλους και γίνεται η μεταφορά αυτών των όπλων. Επίσης ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή της κοινή θέση του 2009. Θα πρέπει να είναι πιο σχολαστικές και δελεχείς εκθέσεις και να δημοσιεύονται ενημερωμένες τακτικά πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο e year old common position is really something unique in the world. Η κοινή θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό είναι κάτι το μοναδικό στον κόσμο και έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, η οποία όμως προφανώς δεν επαρκεί. Το γεγονός είναι πως εμείς είμαστε ο δεύτερος μεγάλος εξαγωγέας, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο. Και αυτό βεβαίως ε, αυξάνεται συνέχεια επειδή μειώνονται οι αμυντικοί προϋπολογισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή μειώνεται και η ζήτηση για όπλα μέσα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν κάνουμε όλο και περισσότερες εξαγωγές. Αφενός λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σαφείς ε, και να γνωρίζουμε πλήρως πού πηγαίνουν τα όπλα που εξάγουμε, γιατί στο σημείο αυτό δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν για να το ξεπεράσουμε αυτό ε, να ενισχύσουμε την κοινή θέση που έχουμε στα πλαίσια της και να ξέρετε πως οι εξαγωγές μεν των κρατών μελών έχουν γίνει πιο ε, διάφανες, αλλά δεν είναι πλήρη τα στοιχεία που δηλώνονται. Πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζεται στην πράξη η κοινή θέση και πώς περνάει μέσα από τα συστήματα των κρατών μελών. Να δούμε ποια είναι η δυνατότητα που έχουμε για να αξιολογήσουμε τον έλεγχο των εξαγωγών ε, των όπλων και ξέρω πως η τελική ευθύνη βαρύνει τα κράτη-μέλη για τη χορήγηση των εξαγωγικών αδειών ή όχι. Ο κύριος Κούκεν έχει το λόγο, μια και ο κύριος Αρλάτσι δεν είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Η σημασία ε, τη Συμφωνίας των Εθνών για το εμπόριο όπλων ε, είναι σημαντική και πιστεύω ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια λογοδοσία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές όπλων. Ιδίως από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από του σημαντικότερους εξαγωγείς όπλων. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη να διασφαλίσουμε τα όπλα να μην συνεισφέρουν σε μεγαλύτερη περιφερειακή αστάθεια, ούτε να εντείνουν εσωτερικές συγκρούσεις. Καταλαβαίνω ότι ενίοτε απεδείχθη δύσκολο για τα κράτη-μέλη να ε, τηρήσουν ε, την κοινή θέση του Συμβουλίου λόγω των διαφορετικών ερμηνεών αυτής. Αυτό αφορά κυρίως το κριτήριο υπερθμών 4, το οποίο ξεκάθαρα προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αρνούνται τη χορήγηση άδεια εξαγωγής αν υπάρχει κίνδυνο στα όπλα να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους από αυτόν της ε, άμυνας. Ε, ή αν υπάρχει κίνδυνος ε, να υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στη σταθερότητα της περιοχής λόγω των όπλων αυτών. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δημόσια διαφάνεια στις εξαγωγές όπλων από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ε, υποβάλλονται εκθέσεις, δημόσιες εκθέσεις. Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο η πολιτική εξαγωγής όπλων, διότι θα μπορούσαν να ενισχυθούν αντί αυτές άλλες πτυχές, όπως είναι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της περιφερειακής σταθερότητας. Πρώτον όμως, και για να έχουμε μεγαλύτερη νομιμοποίηση σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές όπλων, σημαντικό θα είναι τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυστηρά την κοινή θέση του Συμβουλίου. Επίσης θα πρέπει να επικυρώσουν τη συνθήκη περί εμπορίου όπλων. Λίγα βέβαια σημαίνουν τα λόγια που είναι γραμμένα πάνω σε ένα χαρτί. Το σημαντικό είναι να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούκαν. Ο κύριος Χάουι τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Πρόεδρε. Ε, ξέρετε ότι γίνονται ε, πράγματα και θα αυτή τη στιγμή στο Κάιρο και σίγουρα δεν θα πρέπει η συζήτηση μόνο να γίνεται για το πού πάνε σήμερα τα όπλα που εξάγονται που αλλα και σε ποια χέρια μπορούν να καταλήξουν αύριο. Είναι σημαντικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ΜΚΒΟ όπως της Oxfam ε, και της Διεθνούς Αμνηστίας ε, για την συνθήκη αυτή. Ελπίζω η Βουλγαρία να επικυρώσει σύντομα. Η Ισπανία πρέπει να τηρήσει τις διατάξεις όλες οι χώρες πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Η και το Ιράν ήταν οι μόνε χώρε που ήταν κατά ε, συνθήκη. Άρα βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη ακολουθεί τη σωστή πορεία. Εμείς ε, θέλουμε να στηρίξουμε τον κώδικα διοντολογία. Ε, θα πρέπει να δούμε όμως τι θα γίνει και με την αναθεώρηση της κοινή θέσης. Λέτε ότι και με των πολιτών ενημερωμένοι για την αναθεώρηση αλλά μόνο έξι μήνες κράτησαν οι συναντήσεις με τις ΜΚΟ, άρα δεν είναι ε, λογικό αυτό. Πιστεύω ότι όσο θα προχωράει ένα θέρο θα πρέπει να γίνονται όλο και περισσότερες διαβουλεύσεις. Για τα κριτήρια 7 και 8 τώρα, πώς μπορεί η Προεδρία να μα πει ότι δεν υπάρχει καμία καθοδήγηση για τα κριτήρια περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρότι στο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα τη Βαρόνη Άστον γίνεται ειδική αναφορά και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το θέμα στην αναθεώρηση. Μιλάτε για τις ε, ε, ρήτρες διαφάνειας. Ε, θα πρέπει η πρόταση περί δεδομένων να προωθηθεί το Εργατικό Κόμμα ε, έχει προτείνει και αυτό ε, διατάξεις ε, για τον έλεγχο των εξαγωγών. Η Ολλανδία όμως θα έπρεπε και αυτή να κάνει κάτι παραπάνω. Επίσης για την Τσεχία θα ξέρετε 50.000 ε, πιστόλια πολίθηκαν ε, στην Οικητική Αστυνομία του τελευταίου μήνε. Ε, ελπίζω να μην χρησιμοποιηθούν είτε σήμερα είτε τι επόμενε μέρε κατά τρόπο που θα μα κάνει να λυπηθούμε πάρα πολύ για αυτό το γεγονό. Ευχαριστώ, έχετε δίκιο, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Πρέτε για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. το, η βιομηχανία όπλων ε, έχει στρατηγική σημασία σε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πολλά κράτη-μέλη αντιπροσωπεύει μια πηγή μόνιμων εσόδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα όπλων στον κόσμο μετά τη ΣΥΠΑ και ο στρατηγικός χαρακτήρας ε, δεν δικαιολογεί την έλλειψη διαφάνειας. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη ε, την, ε, τα κοινά πρότυπα αναφορά σε ό,τι αφορά τα θέματα της αδειοδότησης. Επίσης θα πρέπει να μας απασχολεί ο προορισμός των εξαγόμενων όπλων. Όταν μιλάμε για εξαγωγές όπλων θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο τελικός προορισμός των όπλων. Οι άδειε ε, μπορεί να εκδίδονται για κάποια κράτη, αλλά εν συνεχεία γίνεται εμπόριο αυτών των όπλων σε άλλες χώρες και τροφοδοτούνται οι τοπικές συγκρούσεις με τον τρόπο αυτό. Τα νομίμως εξαγόμενα όπλα δηλαδή μπορούν να φτάσουν στα χέρια ολοκληρωτικών καθεστώτων και να χρησιμοποιηθούν ε, επομένως για να ε, τερματίσουν τις διαμαρτυρίες της διαδηλώσης του κόσμου. Και βέβαια και να προσέξουμε πολύ και το στρομοκράτς μπορεί να βάλουν χέρι σε αυτά τα όπλα. Η υπογραφή της συνθήκης πιστεύω πάντως ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο έλεγχο και θα βελτιώσει τη διαφάνεια σε αυτό το πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πολλά κράτη-μέλη υπέγραψαν ε, την εν λόγω συνθήκη και εξ αυτών τα 26 είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω και τα δύο να μένα τα κράτη μέλη της Ένωσης να ακολουθήσουν το παράδειγμα των κρατών μελών που ήδη υπέγραψαν και να υπογράψουν και αυτά. Θα πρέπει όλες τις πτυχές που αναφέρθηκαν να τις λάβουμε υπόψη σε ό,τι αφορά το εμπόριο. Ξέρω ότι έχουν γίνει προσπάθειες για την επίλυση. Διακόπτε. Το κύριο Τούσα τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. για τις εξαγωγές όπλων σε τρίτες χώρες είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υπεριαλιστική στρατηγική τις επεμβάσεις και τους πολέμους της ευρωπαϊκής ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της σε διεθνή κλίμακα για τη διασφάλιση της κερδοφορίας και της εξουσίας των μονοπωλίων. χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επέμβαση της ευρωπαϊκής ένωσης και των συμμάχων της στη συρία. σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας telegraph φορτία 3.500 χιλιάδων τόνων όπλων έχουν μεταφερθεί διαμέσου λιμανιών και αεροδρομίων της κροατίας στους σύριους αντικαθεστωτικούς. έτσι την ώρα που ήταν σε εξέλιξη την 1η ιούλη δύο χιλιάδες οι φιέστες για την ένταξη της κροατίας στην ευρωπαϊκή ένωση οι υποδομές και το έδαφος αυτής της χώρας αξιοποιήθηκαν για τους εξοπλισμούς των σύριων αντικαθεστωτικών. ρωτάμε το συμβούλιο και την επιτροπή μετά την απαράδεκτη αυτή απόφαση για την κατάργηση του εμπάρκου όπλων στους αντικαταστατικούς στις 27 του Μάη. Ποια κράτη μέλη εφοδιάζουν, εξοπλίζουν με όπλα τους αντικαταστατικούς στη Συρία. Merci, monsieur Toussas. Et je donne pour terminer la parole à monsieur Leskevicius pour le Conseil. του Συμβουλίου κ. Λεσκεβίτσιος. Νομίζω ότι είπατε εκπρόσωπος ε, σα έχει επιφορτήσει με το να δώσετε εσεί την απάντηση. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, πράγματι, πράγματι εκπροσωπώ. Την είπατε εκπρόσωπο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, διατύπωσαν σχόλια και συστάσεις με βέβαιος ότι θα ληφθούν υπόψη ε, στις συζητήσεις. Υπάρχει ε, μια ομάδα εργασίας όπως γνωρίζετε και σίγουρα όλα όσα ακούστηκαν εδώ θα βοηθήσουν τους συναδέλφους μας και ε, στο στάδιο της αναθεώρησης της όλης αυτής της διαδικασίας. Τώρα απαντώντας Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Χάουιτ και να πω ότι τα κριτήρια 7 και 8 είναι αποτέλεσμα ε, διαβουλεύσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το κριτήριο 2 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και εδώ έχουμε προχωρήσει σημαντικά σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές. Αλλά θέλω να πω ότι η κοινή θέση, νομίζω ότι πολλοί συμφωνήσατε από αυτού, έχει συμβάλει τα μάλα στη βελτίωση του ελέγχου ε, του εμπορίου από τα κράτη-μέλη. Ε, από τα κράτη-μέλη, Υπάρχει μεγαλύτερη υπευθυνότητα, διαφάνεια, λογοδοσία. Η σημερινή συζήτηση αποτελεί μια ακόμη απόδειξη του γεγονότο αυτού. Βέβαια, οποιαδήποτε εκτίμηση, αξιολόγηση τη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτά τα οποία απαγορεύει και αυτά που δεν υπαγορεύει η κοινή θέση. Αυτό το οποίο θεσπίζει η κοινή θέση είναι ένα ενιαίο και μοναδικό θα έλεγα πλαίσιο, το οποίο συνίσταται μεταξύ άλλων σε ανταλλαγή σημαντικών και ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Όμως δεν δημιουργεί μία ενιαία αρχαία διοδότηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ε, πρόκειται για τη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Αυτά ε, θα πρέπει να διεξαγάγουν τους απαραίτητους ελέγχους. Η εναρμόνιση προκύπτει από ε, την ανταλλαγή πληροφοριών και από την άσκηση πιέσεων από τους ομοτήμους των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τις αποφάσεις αλλά επειδή έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό μηχανισμό ελέγχου θα μπορούν ε, και να θεωρούνται υπόλογα σε περιπτώσεις ε, που παραβιάζουν ε, τις σωστές διαδικασίες. Θα πρέπει πάντως και να είμαστε υπερήφανοι για τόσα έχουμε πετύχει. Έχουμε δώσει το καλό παράδειγμα για άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι θετικό. Δεν έχουμε μπει στο δεύτερο πλάνο σε διεθνές επίπεδο. Δείχνουμε υπευθυνότητα. Διαδραματίζουν ένα πολύ προοδευτικό ρόλο και σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την διεθνή συνθήκη, τη συνθήκη του, των Ηνωμένων Εθνών. Η ε, συνθήκη η οποία συμφωνήθηκε στη Νέα Υόρκη τον προηγούμενο μήνα είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο. Θα ενισχύσει την ασφάλεια όσων ζουν σε περιοχές ε, ε, με πολύ σύραξη. Επίσης ε, με τη συνθήκη αυτή μπορεί να δημιουργηθεί και ένα ε, πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού. Όλοι οι όπλων και όχι μόνο τα κράτη-μέλη, θα πρέπει πλέον να, να ε, λειτουργούν υπό τους ίδιους και διαφανείς κανόνες. Όλα αυτά θα επηρεάσουν εν τέλει και θα βελτιώσουν το δίκαιο ανταγωνισμό στο πολύ ευαίσθητο αυτό πεδίο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έληξε η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 για το θέμα αυτό. Και τώρα θα συζητήσουμε την ε, έκθεση του κυρίου Βιτάλ Μουρέιρα για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτική